Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Λόγω της καθυστέρησης οι επεξηγήσεις ψήφου δεν θα γίνουν αμέσως μετά, ε, μετά την ψηφοφορία, αλλά κατά το τέλος της σημερινής συζήτησης θα ψηφίσουμε πρώτα την έκθεση Κίρτσου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έχουμε ονομαστική ψηφοφορία που ειδική πλειοψηφία χρειάζεται. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Και περνάμε στην έκθεση Χριστοφόρου. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Πάλι με ονομαστική ψηφοφορία, πάλι με ειδική πλειοψηφία. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Εγκρίθηκε. Και συνεχίζουμε. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Χρυσόγονου όσον αφορά το αίτημα για την άρση της ε, κοινοβουλευτικής ασυλίας ε, ε, Ευρωβουλευτή. Απλή πλειοψηφία χρειάζεται. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και περνάμε στην έκθεση του κυρίου Σβιεύκα όσον αφορά την άρση του κυρίου ή από του Ιβάν Γιακόφτη, ποιοι υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε και περνάμε στην έκθεση Νεγκρέσκου όσον αφορά την χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, ονομαστική πλειοψηφία, ειδική, ο, ε, ψηφοφορία, ειδική πλειοψηφία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίθηκε και περνάμε στην έκθεση Ρέγνερ όσον αφορά την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κύριου Ουστάσκης. Ο κύριος Φερχόφστατ παρακαλώ έχει τον λόγο. Uh, Σας ευχαριστώ για τη συμπάθεια και τις εθαρρύνσεις. Κύριε Πρόεδρε, μετά την εμφατική συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο Σούλτς, μου είπε ότι τώρα πρέπει να πάρω το λόγο και όχι πριν δύο ώρες. Θα ζητήσω να αναπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή η συγκεκριμένη έκθεση. Γιατί, αν διαβάσει κανείς την έκθεση, Υπάρχουν αμφιβολίες για κάποια πάρα πολύ σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τα Wikileaks και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές αμφιβολίες όταν ασχοληθήκαμε με θέματα τέτοιου είδους στο παρελθόν είπαμε ότι ήμασταν υπέρ της άψης της ασυλίας αλλά παρόλα αυτά είπαμε ότι αυτό δεν θα έπρεπε να τον παρεμποδίσει να ασκεί τα βουλευτικά του καθήκοντα και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είχε πάρει μια τέτοιου είδους απόφαση στο παρελθόν. Δεν πρέπει να περιορίζονται οι προσωπικές ελευθερίες του κυρίου Πάσιτς και δεν καταλαβαίνω γιατί ε, οι προσωπικές ελευθερίες που εξετάζουμε σήμερα, του βουλευτή που εξετάζουμε σήμερα, είναι πιο σημαντικές από τις αντίστοιχες του κυρίου Σέβεριν στο παρελθόν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για διαφθορά. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Φρόφστατ. Σύμφωνα με τον κανονισμό υπάρχει δυνατότητα ένας να τοποθετηθεί υπέρ και ένας εναντίον. Ποιος θέλει να επιχειρηματολογήσει υπέρ του αιτήματο. Ο κύριος συνάδελφος Γκόλνης. Παρακαλώ κύριε Γκόλνης. No. Ich Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Φερχώστατ είναι πολιτικός μου αντίπαλος. Όμως θα υποστηρίξω την πρότασή του. Για πάνω από δέκα χρόνια ήμουν μέλος στην, ειδικά, Ειδική Επιτροπή η οποία τότε λεγόταν Επιτροπή Επαλήθευσης Διαπιστευτηρίων κτλ. κτλ. Έχει υπάρξει σωρία νομολογίας θετικής και όταν υπάρχει το λεγόμενο φούμους περσεκουτιώνης ως μη πολιτικής δίωξης ε, όπου υποτίθεται ότι μπορεί να διώκεται κάποιος για πολιτικούς λόγους πρέπει να διατηρηθεί η ασυλία του. Εγώ νομίζω ότι η νομολογία αυτή την σεβαστήκαμε, τη σέβομαι ακόμα και για τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Δυστυχώς βλέπω ότι η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τίνει να ακολουθεί μια διαφορετική αντίληψη ε, ανάμεσα στους βουλευτές τους οποίους θα ονόμαζα mainstream και από την άλλη ε, διατηρεί διαφορετικές πρακτικές για τους λεγόμενους ανορθόδοξους βουλευτές. Σας ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Γκόνης. Ένα λεπτό έχετε κι εσείς, έχετε τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι άλλοι. Και κύριε συνάδελφε είχα ήδη αποφασίσει ότι ο κύριος Γκόνης λοιπόν υποστηρίζει αυτό το αίτημα. Ποιοι θέλουν να τοποθετούν κατά του αιτήματο. Η κυρία συνάδελφος Ρέγνερ παρακαλώ. Ο κύριος Ουσπάσκιτς είχε διεξοδικότατα ευκαιρία να παρουσιάσει την υπόθεσή του και να δικαιολογήσει τα θέματα. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έδειξε μεγάλη κατανόηση και ήταν πολύ προσεκτική όπως και σε άλλες περιπτώσεις άρσης ασυλίας ασχοληθήκαμε ήδη και κατά την τελευταία κοινοβουλευτική θητεία σε σχέση με την έφεση που έχει ασκηθεί κατά της δικαστικής απόφασης. Και τότε πολύ προσεκτικά εξετάσαμε αυτή την περίπτωση στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Γι' αυτό έχει οριμάσει ο χρόνος να ληφθεί αυτή η απόφαση. Έχουμε επί μεγάλο χρονικό διάστημα ασχοληθεί και εξετάσει σε βάθος την υπόθεση και τώρα ήρθε, ορίμασε η στιγμή να ψηφίσουμε για αυτό το θέμα. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Ρέγνερ. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ψηφίζουμε για την επαναπομπή. Ποιοι είναι υπέρ της επαναπομπής λοιπόν. Ποιοι είναι κατά. Από ό,τι μπορώ να δω είναι η πλειοψηφία, αλλά θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά γι' αυτό για να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε το αίτημα αυτό. Λοιπόν, θα αποφασίσουμε τώρα για το αίτημα αυτό κυρία, της κυρίας Ρέγνερ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε η έκθεση λοιπόν και περνάμε στην έκθεση του συναδέλφου κυρίου Ντούντα που αφορά την ε, η των προνομίων και ασυλιών του κυρίου Αλμπερτίνη. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε το αίτημα. Περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Λαντσμπέργη για τη μακροοικονομική βοήθεια συνδρομή στην Ουκρανία. Έχουμε αρκετέ ονομαστικέ ψηφοφορίε. Ξεκινάμε με την τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Αρχικό κείμενο του άρθρου 1 ε, εδαφίου 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Αρχικό κείμενο. Άρθρο 3 εδάφιο 1. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 11. Υπέρ. Τώρα με διανατάσεως των χειρών. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 5 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τώρα η ψηφο η πρόταση της Επιτροπής ε, θα ψηφιστεί. Συγγνώμη όμως, έχουμε την τροπολογία 6 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τώρα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας συναδέλφου Καϊλή που αφορά την ετήσια έκθεση για την φορολογία. Παράγραφος 5. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 37 με προφορική τροποποίηση της κυρίας Καϊλή. Παρακαλώ. Amendment. It's on. So, uh, welcomes the swift implementation of country by country report. Χαιρετίζει τη γρήγορη εφαρμογή της, ε, των εκθέσεων χώρα ανά χώρα και ζητάει από την Κομισιόν ως επόμενο βήμα να εφαρμόσει υποχρεωτικά τη διαδικασία εκθέσεων αναχώρα ε, ε, ξερώντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς όπου υπάρχουν καθώς και σε φορολογικούς παραδείσους και άμεση αναθεώρηση της λογιστικής οδηγίας και διασφάλιση της ελαχιστοποίησης των διοικητικών αχθών. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, γι' αυτό δεν υπάρχουν. Ωραία. Τότε θα ψηφίσουμε την 37 παράγραφο όσα έχει σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. άποχε. Εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχες Νομίζω εγκρίθηκε, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 39. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Παράγραφος 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 62 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Παράγραφος 67 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Θα ελέγξουμε το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε, είναι σαφές. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Είναι ασαφέ το αποτέλεσμα, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Παράγραφος 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Με την ίδια πλειοψηφία απορρίφθηκε. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Αιτιολογική σκέψη M. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τώρα, το ψήφισμα στο σύνολό του, με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Φτάσαμε στο τέλος των ψηφοφοριών. Θέλω όλους να τους ευχαριστήσω θερμά, όμως κατεπηγόντως να ζητήσω, να παρακαλέσω όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν τη συνεδρία στις Ολομέλειες να παραμείνουν. Εκείνοι που δεν το επιθυμούν να αποχωρήσουν γοργά, διότι θα λάβει τον λόγο η κυρία Μογκερίνη τώρα και πρέπει